Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 9 και 3 λεπτά η ώρα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους. Άλλη μια συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Πριν αρχίσουμε τις ψηφοφορίες μας, θα ήθελα να καλωσορίσω τρεις προσκεκλημένους. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει ήδη. Εδώ είναι. Έχουμε τρία μέλη της Ουκρανικής Βουλής που θα ε, περάσουμε μαζί μας μία ώρα σήμερα το πρωί, η κυρία Οξάνα Ζήρουιτ, ο κύριος Γέγκορος Ζοπότιεφ και ο κύριος Όλαχ Περέσιο. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Εξωτερικών. We then come to the... Ερχόμαστε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Μαραθώνιος σήμερα το πρωί τουλάχιστον μία ώρα και ένα τέταρτο θα ψηφίζουμε. Θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, παρακαλώ, και ελπίζω να τα διακπεραιώσουμε όλα εγκαίρως. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίζουμε το σημείο 10 προς ένα νέο εμπορικό πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης. Η συγκήτρια κυρία Κάτι Πύρη. Δεν ξέρω, θέλει η συγκήτρια να πει κάτι. Όχι, από ό,τι βλέπω. Ωραία, μπορούμε να προχωρήσουμε κανονικά στις ψηφοφορίες. Αρχίζουμε. Έχετε όλοι κάρτες <clears throat> στα μηχανήματα. Ελπίζω. Λοιπόν, προχωρούμε. Τροπολογία υπαριθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ε, τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Συμβαστική 2. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά που πάμε στην τροπολογία 15, όχι. Όχι, έχει καλυφθεί στη συμβαστική τρία. Πού πρέπει να πάμε. On my list, it's... We go... Στο δικό μου κατάλογο λέει τροπολογία 15 τμήμα πρώτο. Όχι, έχει καλυφθεί. <clears throat> Μάλιστα. Άρα. Όχι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 15-1. 15-2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον χρειάζεται έλεγχο αυτό. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Τώρα. Εγκρίνεται.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 εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε, ψήφι υπέρ. Α, όχι, όχι, ηλεκτρονική διορθώνει ο Πρόεδρος, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια κυρία Πύρη. Προχωρούμε τώρα στο Μαυροβούνιο. Που είναι το επόμενο θέμα. Έκθεση σχετικά με την έκθεση Επιτροπής για το Μαυροβούνιο για το 2016. Η συγγετής είναι ο κύριο Στάνοκ. Θέλει να πει τίποτα. Όχι, ευχαριστώ Στάνοκ. Μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν την ψηφοφορία μας. Συμβαστική 2. Ψηφίπε, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 51. Ψηφίπερ. Κατά. Απόχες. Έλεγχος. Παρακαλώ, αρχίζει τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 52. Ψηφιπέ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 4 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 77 τώρα. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 είπε. κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 είπε. κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 96 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ελέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 10. Ορίστε, έλεγχο θέλετε. Μάλιστα, για την 104 ελέγχουμε ηλεκτρονικά αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 επε κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 135 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 147 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Παρακαλώ, ψηφίζουμε την 159 ηλεκτρονικά τώρα, παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα που πάμε. 160. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 161 τσεκ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Δύο κοιμάστε ακόμα. Πέρας. Εγκρίνεται με μικρή διαφορά. 162 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 165 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Αποχές, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, απορρίπτεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές, Ας την ελέγξουμε παρακαλώ. Την 166 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ένας. Εγκρίνεται. 30-27. Ερχόμαστε στον κύριο Κοβάτσεφ, 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 176. Τσόφκο που μόλις κατέφθασε. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Επαληθεύουμε την 179 παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Vote closed. 30 to 28. 30-28 εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. 192. Με προφορική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. 193 σε δύο τμήματα, υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. Στο δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Κυρίου Χατζηγεωργίου, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 7 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 9 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 10 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. Ελέγχουμε παρακαλώ την τροπολογία 10. 59 Απορρίπτεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Απόχες. Έλεγχος. Για την 11. The vote is open. Αρχή η ψηφοφορία. Ένα συνάδελφο δεν ψηφίζει, έχει αποκοιμηθεί. Πέρας 31-27 εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά Παρακαλώ. Κάτι λέει ο κύριος Φλέκενστάιν εκτός μικροφώνου. Ζητήσατε να ελεγχθεί 14. Εχθές. Πότε το ζητήσατε. Ε, τροπολογία 14, λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση του κυρίου Ανδρουλάκη και της κυρίας Ντότς. Ε, ε, ελέγχουμε, αρχίζει ψηφοφορία. Κύριε Φλέκερστάιν, με μπερδεύετε πρωινιάτικα. Πέρασε. Ορίστε. Ήταν προφανές, μου φαίνεται, έτσι δεν είναι. So, we now... Πού είμαστε τώρα. Συμβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ Α, όχι, καταπίπτει, λέει ο πρόεδρος, γιατί εγκρίθηκε 22, 24. Εξαιρετική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Καταπληκτική ψηφοφορία. 25 υπέρ. Κατά. Απόχες. Έλεγχος, παρακαλώ, για την 25. Αρχίζει η ψηφοφορία. Μας λείπει ένας συνάδελφος, παρακαλώ ξυπνήστε. Πέρας. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα πάμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως τροποποιήθηκε η έκθεση αρχίζει τώρα. One colleague is still not participating. Υπάρχει συνάδελφος που δεν ψηφίζει. Πέρας. 51 υπέρ 6 κατά. Εγκρίνεται η έκθεση αυτή. Συγχαρητήρια κύριε Τάνοκ. Macedonia? We now come to the draft report on the 2016. σχετικά με την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο κύριος Ιβο Βάιγκελ είναι εισηγητής. Θέλει να πει τίποτα ο εισηγητής, όχι. Τροπολογία 14 ψήφι Κατά. Αμποχές. Δεν κρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική 8, ψηφιπέ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. Συμβαστική 9, υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. Η τροπολογία 95, ψηφιπέ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. Ερχόμαστε στη συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ερχόμαστε στη συμβιβαστική 13 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στο πρώτο τμήμα της 161. Είναι κατά τμήματα αυτή η ψηφοφορία υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές Ας το αλλάξουμε. Αρχής ψηφοφορία στην 161 τμημα πρώτων. πρώτον. Πέρας. 35-25 γκρίνεται. We then come to the second part who... Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 183 το πρώτο τμήμα της τοπολογίας του κ. Κοβάτσεφ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στη συμβαστική 21 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Παρακαλώ, επαληθεύουμε τη 213. Κοβάτσεφ. προφορία. Πέρασε. 36-24 εγκρίνεται. Συμβιβαστική όχι, προηγουμένως έχουμε πάλι το κύριο Κοβάτσεφ τη 2.14 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.15 Κοβάτσεφ υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εδώ χρειάζεται παλήτευση. Παρακαλώ στη 2.15 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 23 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη 228. Κατά τμήματα. Ο έχει ζητήσει ο εισηγητής ο ίδιος. Τμήμα πρώτον ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 233 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβαστική 24 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.45 είπε, Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.48 είπε, Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.49 είπέ, Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.50 υπέρ. Κατά αποχές Ας επαληθεύσουμε τη 250 παρακαλώ. Κύριε Καστάλτο, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε, εγκρίθηκε. 2.51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.53 υπέρ, κατά, αποχές ε, ε, έλεγχος στη 253 παρακαλώ επαληθεύουμε αρχίζει η ψηφοφορία The vote Απορρίπτεται. Η 254 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 συμβιβαστική ψήφη. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 259 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίφτεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στη συμβαστική 27 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα που πάμε, 2.83 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στο δεύτερο τμήμα της 300 μάλλον, εφόσον εγκρίνονται όλα αυτά, γιατί βρω κιόλας. Πού είναι 300. Στο δεύτερο τμήμα ήδη. Μάλιστα. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 301. Σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 304 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 315 υπέρ. Κατά. Αποχές Ας την ελέγξουμε παρακαλώ την 315 αρχίζει η επαλήθευση. Πέρας. Wow. Μάλιστα. Ήταν προφανέστατο. Ποια ήταν αυτή. 3.15. Λοιπόν, προχωρούμε. 3.16 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 3.18 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 27, ψήφι υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές έλεγχος. 27 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 28 είπε, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 είπε, Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Την 29. Επαληθεύουμε αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Μας λείπουν 3, 2, Ποιο λέει, κύριο Φλέκενστάιν, μακάρι να Λοιπόν, πέρα εγκρίθηκε. Η 30 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίθηκε. 37 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική, μάλλον όχι, 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ το πρώτο τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος το δεύτερο τμήμα της τοπολογίας 55 Ένας απερίφθη με δύο ψήφους διαφορά 29-31 συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία 8. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές την ελέγχουμε αυτή. Τη 10 παρακαλώ αρχίζει η επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίθηκε. 11 και 12 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται η 13 υπέρ κατά αποχές έλεγχος στη 13 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίθηκε λοιπόν τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική για το σύνολο του σχεδίου έκθεση όπως τροποποιήθηκε, αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίθηκε. 54 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. You tell me this one. Ah, Περνάμε στο επόμενο θέμα της τη σχετικά με την έκθεση Επιτροπής της Σερβία του 2016. Θέλει να πει κάτι ο συγγετής. Όχι, αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζουμε με την ε, πρώτη ε, συμβαστική τροπολογία. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερη υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72. Μπόγκοβιτς Κουκάν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 83. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται η 83. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Στην ε, σελίδα 5 του εγγράφου ψηφοφοριών. Λούνατσεκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 174. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 175. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 176. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθεια στην 176. Εντάξει. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 177. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 181 Καστάλτο Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με σαφή πλειοψηφία. Συμβιβαστική 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 228 αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 2.29 υπέρ κατά αποχές Από την αριστερή πλευρά δεν είδα και μεγάλη συμμετοχή, την επαναλαμβάνουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 229. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 230 υπέρ κατά αποχές Πάλι το ίδιο πρόβλημα. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν της 230. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 243. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 244. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 245. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 246. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 247. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 249 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.51 2.52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 2.53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 2.54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για 293 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 294 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 295 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 308 Τάνοκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 323 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 325 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φάνουμε τώρα στις επόμενη σειρά τροπολογιών. 17 υπέρ κατά ε, αποχές 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 19 υπέρ κατά αποχές συγχαρητήρια, 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 23 υπέρ κατά Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 23. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση θέλετε. Εντάξει. 24. Αρχίζει ψηφοφορία. Τρεις συνάδελφοι. Ε, εντάξει, ψήφισαν με καθυστέρηση. Έχει καλώς, εγκρίνεται. 25. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 29 αρχίζει ψηφοφορία Λείπει κάποιος. Τέλος πάντων. 28 προς 33 απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά αποχές 31. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 32. Με συγχωρείτε, απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε on block από το 1 έως το 10 τον, της, τον κύριο Βιλιμσκι υπέρ κατά αποχές. Απερίφθησαν όλοι. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φτάνουμε τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία της έκθεσης έτσι όπως την τροποποιήσαμε. Το σύνολό της αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται με 55 προς 2. Πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Φτάνουμε τώρα στο επόμενο, επόμενη έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του Κωσυχοπέριου του 2016. Θέλει να πει κάτι η συγγήτρια, όχι, ο κύριος Παντζέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι οι σοσιαλιστές δεν θα ψηφίσουν την συμβιβαστική τροπολογία 4 δεδομένου ότι δεν ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις των τίνων εκθέσεων που θα πρέπει να δίδουν μια πιο λεπτομεριακή εικόνα και όχι μια στιγμή εικόνα του ακριβώς γίνεται. Είπαμε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν το κόσυφο πέδιο. Εδώ πέρα λοιπόν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από πολιτικής πλευράς. Δεν μπορούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν να ψηφίσουμε αυτή την συμβαστική τροπολογία που προανέφερα. Κύριε Παντζέρη. Δεν θα ψηφίσετε την συμβαστική τροπολογία 4, δεν είναι έτσι στους σοσιαλιστές, δεν είναι έτσι. Η κυρία Λούνατσεκ. Θες το μεσημέρι, όταν ήρθα σε επαφή με τους άλλους συναδέλφους, κάτι άλλο μου είπαν οι σοσιαλιστές, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Τώρα ακούω κάτι διαφορετικό. Χθε κάτι από το ΕΛΚ. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, η αρχική μου πρόταση ήταν το Κοινοβούλιο, όπως και στο παρελθόν πολλές φορές, ενθαρρύνει ε, κράτη-μέλη, τα πέντε που δεν έχουν αναγνωστικό να το κάνει. Θα πρέπει λοιπόν και εγώ να βάλω μία σε αυτή τη πρόταση. Θα δούμε στην ψηφοφορία τι θα γίνει. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα πάρουμε ως κάτι θετικό που γίνεται. Το Μπαγκλαντές προχθές ε, ε, ως επίσημη χώρα του. Επίσης αναγνώρισε το Κωσυφοπαίδιο. Τα πέντε λοιπόν εναπομείναν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το κάνουν. Είναι θέμα πρόεδρου και αυτό. Αυτό είναι το σχολείο μου. Δεν υπάρχει άλλο σχόλιο. Θα αρχίσουμε την ψηφοφορία, λέει ο Προεδρεύων. Η συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 και 48. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 49. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση της 50 του κυρίου Αντάκτουξον. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 48 προς 10. Σαφής ε, υιοθέτηση. 51 υπέρ κατά ε, εγκρίνεται. 50, απορρίπτεται 52. Απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοίτα περίφημη. Όχι, όχι, όχι, δεν φτάνουμε ακόμη. Όχι, όχι, λέει ο πρόεδρος. Λάθος, δεν φτάσαμε ακόμη. Σαφχάουζεν Κόρβιν Μίκε, 74-75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 76 και 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 79 και 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 82-83. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Ηλεκτρονική επαλήθευση των 82 και 83. Υπέρ, ε, ανοίγει ψηφοφορία, συγγνώμη. Λίγη ψηφοφορία. Σαφώς. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ κατά αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της συμβιβαστικής 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 27 προς 25. Συμβιβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111. Πάει. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία 3. Λίγη. Η ψηφοφορία 30 προς 31. Απορρίπτεται λοιπόν. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 142. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση 142, αρχίζει ψηφοφορία. Ένας μας λείπει. Ας ψηφίσει. Λίγη ψηφοφορία. 38 προς 22 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 152 πύρη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση 153 Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 154. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές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 Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 197. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 198. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 199. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση 199. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 9 προς 28, 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 205 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση της 205, αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται. 240. 7. Ταμπάσκι, ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη η ψηφοφορία εγκρίνεται. 248 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 249 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 250 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση 250, αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 251 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 252 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 253 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 254 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση 254 αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Κάνουμε, φτάνουμε στη 256. χωρίς Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 257 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 250, ε, εγκρίνεται συγγνώμη, 258 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 200, 200, we just voted. 260 ψηφίσαμε. Α, λέει ο πρόεδρος. Α, προσπαθούσα να δω αν είστε Ξύπνη, ξύπνοι. Τέλος πάντων, 260, την εγκρίναμε, 261. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 269 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 270 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 271, 72 και 73 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 2.74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.78 και 2.79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 2.75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.76 υπέρ κατά αποχές απερίπτεται. 2.80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 287 Ράντος Γιάσκοβιτς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 289 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 292 χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση του δευτέρου μέρους της 292. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 293. Μιλάν μόνο. Υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 και 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση 24 αρχίζει ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 και 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση στις 31. Αρχίζει η ψηφοφορία. All on board, the vote is closed and this has been rejected. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση 32. Αρχίζει ψηφοφορία. This is... Εγκρίνεται με 29 προς 28. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 και 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται μάλλον. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Ε, Με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε ταυτόσιμες τροπολογίες 1 προς 4 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. σαφώς απορρίπτονται αυτές οι τροπολογίες. Και τώρα φτάνουμε στην ε, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία της έκθεσης έτσι όπως την τροποποίησαμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ένα συνάδελφος δεν έχει ψηφίσει ακόμη. Λίγη ψηφοφορία. 40 προς 12 εγκρίθηκε. So, shall we continue? Να συνεχίσουμε. Υπότιτλοι for information Dear colleagues, it's 20 past. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι 10 και 20. Ο κύριος Σόλτς είναι σε άλλη ψηφοφορία για το 15, από ό,τι βλέπω. Μισό λεπτό. 16 is okay. What we will do... Κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Θα εξετάσουμε πρώτα το 16 και μετά το 15. Γιατί η κυρία Μανέσκου είναι εδώ, η συντάκτρια της γνωμοδότησης. Επομένως, περνάμε στο 16, θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκο τρίτης χώρας ή από απάτριδα. Εξετάζουμε τη γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ για την αναδιατύπωση ε, του κανονισμού και η συντάκτρια είναι η κυρία Μανέσκου από το ΕΛΚ. Σύμφωνα με, τους σχετικούς, ε, με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού ε, γίνονται παραδεκτές μόνο οι τροπολογίες επί τμήματων του κανονισμού που αλλάζουν. Η κυρία Μανέσκου έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε συζητούμε ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα και εκφράζουμε εμείς μια γνωμοδότηση, μια άποψη. Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή είναι η ΛΥΜΠΕ, η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών και μας ζητείτε να τροποποιήσουμε ένα κανονισμό που υποτίθεται ότι είναι λύση στο πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα σήμερα, την προσφυγική κρίση. Έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία υπογραμμίζει δύο βασικές πτυχές. Πρώτον, το σκοπό του κανονισμού, δηλαδή να θέσει ένα τέλος στην χαοτική και παράτυπη και παράνομη μεταναστευτική διαδικασία και να αντικατασταθεί με νόμιμους και ασφαλείς ε, δρόμους εισόδου στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια για τους νομίμους ετούντες άσυλου και δεύτερο σκοπό είναι να να αναγνωριστούν και να λυθεί το θέμα αυτών όλοι αυτοί που δεν έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να χαίρουν διεθνούς προστασίας. Ο μόνος τρόπος για να μεταναστεύσει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να ζητήσει τη διεθνή προστασία και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ικανότητα και το μηχανισμό να λύσει τα ζητήματα της παράνομης ή παράτυπης μετανάστευσης με αυτόν τον τρόπο. Συζητώντας τώρα με τους συναδέλφους και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αυτών, καταλήξαμε στο εξής συμπέρασμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν σημειώνει επιτυχίε στην επίλυση αυτού του ζητήματος και σύν τη αλλη καποια κάποια κράτη-μέλη ζητούν ένα μόνιμο σύστημα για το μοίρασμα των βαρών ενώ άλλα κράτη-μέλη θέλουν τη διατήρηση και το streamlining, την ευθυγράμμιση του υφιστάμενου συστήματος. Άρα τα κράτη-μέλη διείστανται, είναι πολύ ε, διαφορετικέ οι θέσει των μεν και των δε. Συμφωνούμε απολύτω ότι είναι προφανές ότι το σημερινό κείμενο έτσι όπως έχει επιδέχεται ουσιαστικών βελτιώσεων και αυτό συμβαίνει διότι οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της θεμελιώδου μεταρρύθμισης του υφιστάμενου συστήματος. Το εφιστάμενο σύστημα βεβαίως δεν ήταν απολύτως τέλειο και δεν ήταν και καθόλου λειτουργικό και όλα αυτά αποδείχθηκαν όταν ξέσπασε η κρίση αυτή. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω τα βασικά προβλήματα του κανονισμού. Πρώτον, ο μηχανισμός αναδιανομής λόγω του αυτόματου χαρακτήρα του μηχανισμού αναδιανομής, ο μηχανισμός αυτός δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και προϋποθέσεις που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος και γι' αυτό θεωρούμε ότι οποιαδήποτε πρόταση για την ανακατανομή ε, των διεθνών διεθνώς ετούντων διεθνούς προστασίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και την ικανότητα υποδοχής του κάθε κράτους μέλους. Για παράδειγμα, το ποσοστό ανεργία θα μπορούσε να είναι μια τέτοια πτυχία, ένα τέτοιο σκέλο. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ποσοστό ανεργία που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό όρο. Και θα είναι δύσκολο για αυτά τα κράτη-μέλη να υποδεχθούν και να δώσουν καταφύγιο σε μετανάστες. Όμως το πρόγραμμα και το σύστημα ανακατανομής ε, για τη μετεγκατάσταση αποδείχθηκε απολύτως δυσλειτουργικό. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το οικονομικό σκέλος. Το δίκαιο μοίρασμα των ευθυνών δεν μπορεί να ξεκινά με τις οικονομικές κυρώσεις έναντι ορισμένων κρατών μελών δύσκολα μπορεί κανείς να καταλάβει και να διανοηθεί πώς θα εφαρμοστεί μια τέτοια διάταξη. Ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούν ότι ο εθελούσιος χαρακτήρας και τα ρεαλιστικά κριτήρια είναι και τα εχέγγυα για την επιτυχή επίλυση αυτού του προβλήματος και οι δευτερογενείς μετακινήσεις βεβαίως. Τρίτη πτυχή είναι τα ειδικά κριτήρια για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης 250.000 ευρώ ανά άτομο και εγώ και η κυρία Βίξτρομ αυτό το συζητήσαμε και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών δυσκολεύεται να δεχθεί αυτό το συγκεκριμένο κριτήριο έτσι όπως προτάθηκε δεν γνωρίζουμε τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν και θα επιβληθούν στα κράτη-μέλη για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης. Τώρα, για τις δευτερογενείς μετακινήσεις, τα εργαλεία που προβλέπει ο κανονισμός δεν είναι αρκετά και δεν είναι επαρκή να σταματήσουν τις δευτερογενείς μετακινήσεις υπηκών τρίτων χωρών. Οι μεταφορές ε, δεν είναι πολύ αποτελεσματικές, οι διαβιβάσεις μάλλον, και δευτερογενή μετακίνηση γίνεται μετά από ατελή μεταφορά. Πέμπτον, το σύστημα το πληροφοριακό που περιέχει λεπτομέρειες για τη ε, θέσπιση και λειτουργία συστημάτων τεχνολογίας και πληροφορικής για την καταχώρηση των ε, δεδομένων ταυτοποίησης. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει σαφή και δεν έχουν διευκρινιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κανονισμός είναι ένα κλειδί ανακατανομής υποχρεωτικό και μόνιμο και δεν λειτουργεί με την διαδικασία ε, του επίγοντος όταν συμβαίνει κάτι επίγον. Μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις λοιπόν θεωρούμε ότι το κείμενο μπορεί να βελτιωθεί. Ε, με βάση τη δική μας οπτική γωνία, την οπτική γωνία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν συζητούμε για ένα πρόβλημα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να υποδέχεται και να έχει ένα σαφή μηχανισμό για την υποδοχή των μεταναστών που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Δεν συζητούμε μόνο αυτό, αλλά συζητούμε και για προβλήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν υπό την αιγίδα, αν θέλετε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Και γι' αυτό είμαστε εδώ παρόντες για να βελτιώσουμε το κείμενο. Περιμένω να συνεργαστώ στενά με τους συναδέλφους, με τους κοιόδης εισηγητές, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προτείνει αυτό το κείμενο. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ήταν πολύ βοηθητική, όμως η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων δεν έχει ακόμα συνταντηθεί με εμά και δεν μας έχει δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Παραμένω όμως στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μανέσκου για την παρουσίαση της νομοδότησης. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Παντζέρη, πρώτος από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με την κυρία Μανέσκου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και ανεπαρκής και ατελής, γιατί δεν υπερβαίνει τα διαστοτικά προβλήματα, τα δομικά προβλήματα του μεταναστευτικού φαινομένου. Εμείς καλούμαστε τώρα να κάνουμε μια δουλειά. Εγώ θα επικεντρωθώ στα εξή τέσσερα σημεία που θεωρώ σημαντικά. Πέντε δηλαδή. Πρώτον, το μηχανισμό ε, κατανομής στην ε, πρόταση. Αυτό που λείπει είναι η αλληλέγγυα προσέγγιση ε, που να κατανέμει ε, σωστά και να επιμερίζει και τις ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής. Τι μας λέει η πρόταση, ότι το Δουβλίνο 4 ε, αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αναλάβουν και να υποδεχθούν κάποιους ετούντες άσυλο. Διότι ο μηχανισμός κινητοποιείται μόνο όταν μια χώρα λάβει δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων. Πρέπει να εισαχθεί εδώ το στοιχείο της αλληλεγγύης. Δεύτερον, τι γίνεται με τις περιπτώσεις ε, απαράδεκτων αιτήσεων. Ε, τα κράτη-μέλη παραμένουν ε, στα σύνορά τους ως μοναδικοί αρμόδιοι να διαχειριστούν και να διεκπαιρεώσουν τις αιτήσει ασύλου. Δηλαδή, αν ετών άσυλο έχει περάσει από τρίτη χώρα, η οποία θεωρείται ασφαλής και έχει ζητήσει άσυλο, έχει ζητήσει προστασία, ε, δεν γίνεται σωστά η ε, κατανομή ε, της γραφειοκρατικής δουλειάς. Και επίσης θα πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε ασφαλή χώρα. Γιατί υπάρχουν και θέματα θρησκευτικών μειονοτήτων. Τρίτον, αναφέρθηκε και η κυρία Μανέσκου στις κυρώσεις. Έχω την εντύπωση ότι αυτό γίνεται με παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί οι κυρώσει είναι κάτι το οποίο έχει εισαχθεί για να προλαμβάνονται καταχρήσεις και δευτερογενείς μετακινήσεις. Όταν κάποιοι ετούνται σε άσυλο, ας πούμε, δεν σέβονται και παραβιάζουν την υποχρέωση που έχουν να παραμένουν στη χώρα στην οποία έχουν ζητήσει για πρώτη φορά άσυλο. και γίνεται λόγος για τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματα υποδοχής και ε, τα δικαιώματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε επίγουσες περιπτώσεις. Υπάρχει και η δυνατότητα έτσι ασύλου στις πρεσβείες. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα, εάν θέλουμε να αποφύγουμε επικίνδυνα ταξίδια ανθρώπων που φεύγουν από σειράξει να έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν σε τρίτες χώρες τις πρεσβείες των κρατών ή ε, στα προξενία ε, αίτηση ασύλου. Άλλο θέμα, προστασία ανηλίκων και ε, ευάλωτων προσώπων και ομάδων. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά να μην υπάρχουν ανακαστικές μετακινήσεις ανηλίκων ε, εις βάρος των δικών τους ε, σύμφερων. Θα κάνουμε τροπολογίες και ελπίζουμε να βοηθήσουν. Ευχαριστώ. Next speaker. Ευχαριστώ. Από την άλλη, κυρία Βόλτμαντς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι από το 2014 αντιμετωπίζει η Ευρώπη μια άνευ προηγουμένου μεταναστευτική κρίση. Το 2015 1.260.000 άνθρωποι υπέβαλαν αίτημα διεθνούς προστασίας στα 28 κράτη-μέλη. Και πέρσι 1.175.000 άνθρωποι υπέβαλαν τέτοιο αίτημα. Οι επικεφαλείς, οι κρατών και κυβερνήσεων φέρουν τεράστια ευθύνη. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν τη διαχειρίστηκαν σωστά αυτή την κρίση, δεν την προέβλεψαν, δεν οργάνωσαν, δεν ρύθμισαν σωστά τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Αυτό το χάος, αυτή η ανοργανωσιά είναι αυτό που έχει γεννήσει το φόβο στα κράτη-μέλη. Αυτή η έλλειψη συνολική πολιτική διαχείρισης έκανε κάθε χώρα εσωστρεφή, στραμμένη προ τον εαυτό της και εκφράζω τη βαθιά μου λύπη γι' αυτό. Η Ευρώπη ε, ουσιαστικά ε, σπατάλησε χρόνο Είναι επίγον να εναρμονίσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα ασύλου. Θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταρρυθμίσει το Δουβλίνο, να προβλέψει ασφαλείς διόδους μεταφοράς, μετάβασης για τους πρόσφυγες από τη Συρία και να δείξει αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα. Και η πρόταση μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να επιδείξει μεγαλύτερο βάρος και φιλοδοξία, κυρίως σε δύο επίπεδα, τα οποία θέλω να σας αναφέρω, καλό, παρόλο που δεν εντάσσονται απολύτως στο πεδίο αρμαδιότητας της Επιτροπής μας. Ως προς το μηχανισμό μετεγκατάστασης, αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ιταλία και στην Ελλάδα, είναι κάτι που μας αφορά όλους εμάς και όχι μόνο αυτές τις δύο χώρες. Η τεράστια πλειοψηφία μεταναστών και προσφύγων φτάνουν σε αυτές τις χώρες, στην Ιταλία και την Ελλάδα, απλά και μόνο για γεωγραφικούς λόγους, επειδή αυτές οι χώρες βρίσκονται στις θύρες της Ευρώπης Ευρώπης. Δεύτερον, κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως, η ασυνόδευτοι ανήλικοι. Η κατάσταση έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή πρέπει να βελτιωθεί με συγκεκριμένα, στοχευμένα μέτρα. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μας μεταχειρίζονται αυτά τα παιδιά ε, μην ε, μεριμνώντας καθόλου ε, για τις διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού, για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια αυτών των παιδιών. Πήγα στη Δουνκέρκη την περασμένη εβδομάδα και αυτά που είδα εκεί πρέπει να σας πω με πάσα ειλικρίνεια, είναι αποτρόπια. Εάν εγώ μεταχειριστώ στην πατρίδα μου το σκύλο μου με τον τρόπο με τον οποίο οι Γάλλοι μεταχειρίζονται αυτά τα παιδιά στη Δουκέρκη, σίγουρα θα έρθει η ένομη τάξη και θα μου πει στην πατρίδα μου αυτό δεν είναι αποδεκτό και θα με τιμωρήσει. Πηγαίνετε κύριε Πρόεδρε να το δείτε, δεν θα πιστεύετε τα μάτια σας. Είναι επίσημο γαλλικό ε, στρατόπεδο, ε, επίσημος γαλλικός καταβλισμός προσφύγων και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας γιατί αυτά που είδα εκεί είναι φρικτά. Ε, στηρίζω τη συνάδελφο κυρία Μανέσκου. Θα προτείνω κάποιε τροπολογίε ωστόσο για να ενισχυθεί η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίω ε, σε ό,τι αφορά τι νόμιμε οδού πρόσβαση προσφύγων και μεταναστών που χρήζουν διεθνού προστασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βαλέρο από τους πράσινου παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ενδεχομένως χρειάζεται να αλλάξει το Δουβλίνο. Είναι κάτι που το έχουμε πει επανειλημμένος. Ποτέ δεν δούλεψε. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε αυτή τη τεράστια ροή ε, προσφύγων και μεταναστών προς την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, το να ε, μιλάει κανείς ε, για μοίρασμα βαρών. Ε, δεν μπορεί κανείς να μοιράσει βάρη χωρίς να είναι εθελούσιος ο χαρακτήρας. Πρέπει να μοιραστούν οι ευθύνες. Δεν μου αρέσει η λέξη το μοίρασμα των βαρών. Ε, πρέπει να αναλάβουμε από κοινού τις ευθύνες. Εμείς πρέπει οι ίδιοι να αυτοπεριοριστούμε και να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη και να ασχοληθούμε με θέματα ασύλου από κοινού. Να μην μιλούμε για ένα βάρος το οποίο θα πρέπει να μοιραστεί, αλλά για μια ευθύνη που θα πρέπει να αναλυφθεί. Ας μην μιλήσουμε λοιπόν για μοίρασμα βαρών, ας μιλήσουμε για ε, από κοινού ανάληψη ευθυνών. Πρέπει να αλλάξει και η γλώσσα και η διατύπωση για να αλλάξουν και οι νοτροπίες. Οφείλουμε να έχουμε τα κατάλληλα συστήματα ελέγχου των ετούντων άσυλο. Είναι μεγάλο το πρόβλημα σήμερα και δεν έχουν όλες οι χώρες τα κατάλληλα συστήματα ε, για τον έλεγχο και την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου. Δεν ξέρω πόσο θα διαμορφωθούν όλα αυτά και πώς θα συνδυαστούν με την υπόλοιπη δουλειά που κάνουμε εμείς στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με πράγματα που γίνονται εντός Ευρώπης, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και λιγότερο έχουν να κάνουν με αυτό που γίνεται εκτός Ευρώπης. Όμως, όπως το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προτάσεις που τίθενται επιτάπητος για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Προσπαθούμε να πείσουμε το Συμβούλιο ότι χρειάζεται και η ανθρωπιστική θεώρηση, η βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να διασχίσουν τη Μεσόγειο ε, οι άνθρωποι αυτοί, αλλά να υποβάλουν το αίτημά τους σε αντίστοιχη ευρωπαϊκή ε, πρεσβεία ε, που βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκών συνόρων. Δεν είμαστε σίγουροι βέβαια ποιες είναι οι ασφαλείς χώρες και αυτή η σύνδεση είναι κάπως δύσκολη. Πιστεύω όμως ότι μπορεί να γίνει. Οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας τη διαφορά μεταξύ οικονομικού μετανάστη και τούντα άσυλου. Άσυλο. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν και τις δύο αυτές ιδιότητες και όταν ε, εξετάζουμε ένα φάκελο βλέπουμε ένα νεαρό Αφγανό ή μια νεαρή Αφγανή για παράδειγμα που φτάνουν εδώ και που θεωρούνται οικονομικοί μετανάστες. Ωστόσο, στο τέλος της διαδικασίας, ακριβώς επειδή θεωρούνται οικονομικοί οι μετανάστες, στέλνονται πίσω στην πατρίδα τους. Ενδεχομένως μέσω μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας όπως η Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι κατά πόσο είναι σωστή αυτή η διαδικασία. Τι κάνουμε με τους ανθρώπους που στέλνονται πίσω. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά άπτονται και του πεδίου αρμοδιότητας της δικής μας Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και γι' αυτό θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες που μας αφορούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Επιτίδιος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τρόπος αντιμετωπίσεως των ε, κυμάτων, των ε, νομίμων και παρανόμων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο τρόπος και ο μηχανισμός χορηγήσεως ασύλου ε, δεν είναι αποτελεσματικός και λειτουργικό. Πρέπει όμως να κάνουμε κάποιες διακρίσεις, ούτω ώστε να διευκολύνουμε τις προσπάθειες και χορηγήσεω ασύλου, αλλά κυρίως αντιμετωπίσεω του κύματο των παρανόμων μεταναστών. Δεν μπορούμε να χορηγούμε άσυλο σε όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες οι οποίοι έρχονται κατά κύματα κυρίως στις ε, χώρες των εξωτερικών συνόρων, την Ελλάδα και την Ιταλία, διότι έτσι καταργούμε ουσιαστικά και καταστρατηγούμε την έννοια του ασύλου. Άσυλο πρέπει να λαμβάνουν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη, διώκονται και υπάρχει ενδεχόμενο, εάν επιστρέψουν στην πατρίδα τους, να υποστούν βασανιστήρια, ακόμη και το θάνατο. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους, να υπάρχει μια αλληλεγγύη όλων των κρατών, κυρίως προς τα κράτη των εξωτερικών συνόρων, διότι δεν είναι δυνατόν όλοι όσοι ζητούν άσυλο να, πάρουν, λάβουν άσυλο είτε στην Ιταλία είτε στην Ελλάδα. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Να γίνει η κατανομή αυτών που ζητούν άσυλο αλλά και των ε, μεταναστών και των προσφύγων κατά τρόπο δίκαιο σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να θέλουμε να κάνουμε πολιτική και, να, και κάποια κράτη να κάνουν τον καλό Σαμαρίτη και από την άλλη μεριά να μην δέχονται μετανάστες ή πρόσφυγες στην επικράτειά τους. Και τέλος, ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και σοβαρά υπόψη είναι να μην επιστρέφουν όποτε θέλουν τα κράτη αυτά τα οποία χορηγούν άσυλο σε κάποιους ή παίρνουν κάποιους ε, μετανάστες ή πρόσφυγες στην επικράτειά τους να τα στέλνουν πάλι στα κράτη της πρώτης ε, εισόδου. Αυτό και δίκαιο δεν είναι και δυσλειτουργικό και εν πάση περιπτώσει δεν συμβάλλει στην ε, συνεργασία και τη δημιουργία κλίματος αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank Any further? Στο. Οπότε, να θυμίσω λίγο το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία κατάσταση τροπολογιών, 3η Μαρτίου. Εδώ στην Επίτροπή μας, μάλλον θα ψηφίσουμε στις 10 και 11 Απριλίου. Ωραία. Να επανέλθουμε στο σημείο 15 ο κύριος Σόλτς, εισηγητής, κατέφθασε. Αυξάνονται οι σχέσεις μας και συσφίγουμε τις σχέσεις με την Μογγολία. Ε, είναι δημοκρατική χώρα, σπάνιο πράγμα για την περιοχή. Συμφωνήσαμε μια ε, το 2013 εταιρική σχέση και συνεργασίας. Την περασμένη εβδομάδα έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του το Κοινοβούλιο με, με ένα συνολικό ψήφισμα για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Μογγολίας. Σήμερα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για ένα συμπληρωματικό πρωτόκολλο για ένταξη και της Κροατίας στη Συμφωνία εταιρική Σχέσης και Συνεργασίας. Χρειάζεται και κύρωση. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Χέλμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και για την κατανόηση γιατί ψηφίζουμε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, γι' αυτό καθυστέρησα. Ε, τώρα μόλις μπορώ να σας μιλήσω για το θέμα αυτό. Δεν έχω να προσθέσω πολλά περισσότερα σε σχέση με όσα είπατε εσείς, Πρόεδρε. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής και της τοποθέτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στην περισμένη σύνοδο του Στρασβούργου για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, τώρα χρειάζεται και σύμφωνη γνώμη σχετικά ε, με την συμπεριψή και της Κροατίας στο συγκεκριμένο ε, πρωτόκολλο και συμφωνία. Θα συνιστούσα λοιπόν στην Επιτροπή Εξωτερικών και σε όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας και για τη διαδικασία αυτή βασιζόμενη στο σχέδιο θέσεως του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς από καμιά άλλη πολιτική ομάδα θέλει να πει τίποτα για το συγκεκριμένο θέμα. Not the case. Όχι, από ό,τι βλέπω, κανείς από τους κοιόδης. Οπότε, έχουμε προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 3 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι, ενώ η ψηφοφορία εδώ θα γίνει 20 και 21 Μαρτίου, ε, μία από τις δύο μέρες, ενώ για την Ολομέλη έχει προγραμματιστεί για τη σύνοδο του Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και φτάσαμε στο σημείο 17. δημοσιονομική κανόνες που εφαρμόζεται στο Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης στην αναθεώρηση ε, των γενικών ε, διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού με άλλα λόγια Βέβαια το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο και πάρα πολύ τεχνικό, αλλά πολύ σημαντικό και για μας, διότι πολύ συχνά τα οικονομικά καθορίζουν ε, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, ως γενική παρατήρηση έχω να πω ότι οι γενικοί κανόνες ε, πλέον είναι απλούστευση και η ορατότητα. Θέλω να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Κριστέα, για να μα παρουσιάσει. Δεν σα έβλεπα και τη γνωμοδότηση. Παρακαλώ, κύριε Κριστέα. Um, now, for the spectrum of... Για την ΑΦΕΤ, είναι περιορισμένο το φάσμα της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, αλλά έχετε δίκιο να λέτε ότι παρόλα αυτά είναι κρίσιμο, γιατί οι αλλαγή στους δημοσιονομικούς κανόνες άμεσα επηρεάζουν και την αποτελεσματικότητα και την γενικότερη δράση μας στα εξωτερικά. η γενική στόχη είναι συνοχή, απλούστευση των οικονομικών κανόνων και αυξημένη ε, ευελιξία στη διαχείριση του προπολογισμού. Αν δούμε την πρόταση από μια γενική σκοπιά, οι προτεραιότητες αυτές προφανώς μας βρίσκουν σύμφωνους. Πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε για το γεγονός ότι χρειάζεται απλούστευση των κανόνων και η διαχείριση του προπολογισμού ταυτόχρονα να γίνει πιο ευέλικτη. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις εξωτερικές σχέσεις. Αλλά η ευελιξία και η απλοποίηση δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των αρχών και αξιών πρώτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά δεύτερο λόγο και κατά τρίτο των βασικών στόχων των σημερινών ε, εργαλείων και μέσων ε, χρηματοδοτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, στα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς και τι έχει πολιτική σημασία πρέπει να παρακολουθούμε και να προσέχουμε. Πρώτον, υπάρχει ένα συγκεκριμένος τομέας που αφορά τα ε, χρηματοδοτικά μέσα ECI, ΕΠΑ, ΕΝΗ που αφορούν ε, εξωτερικές δράσεις. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μαξιλαράκι ε, ευελιξίας. Υπάρχει ο κίνδυνος. Γιατί ένα 10% ε, των κονδυλίων αυτών ε, παραμένουν αδιάθετα και υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθούν αυτές οι πιστώσεις. Το θέμα λοιπόν είναι πώς ε, διατίθενται και με ποιο τρόπο καθορίζεται. Το άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι τα καταπιστευματικά ταμεία. Υπάρχει θέμα διαφάνειας και λογοδοσίας. Τα ταμεία αυτά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουν την προστιθέμενη αξία τους, αλλά έχουν και κάποια ερωτηματικά, ε, όπως είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τέλος, ε, είδαμε και τι γίνεται με τις δημόσιες προμήθειες και συμβάσεις στην εξωτερική δράση. Ε, στο κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας χρειάζονται κάποιες διαδικαστικές αλλαγές και είναι και το πνεύμα των αλλαγών που προτείνουμε εμείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά ήταν όλα όσα ήθελα να πω. Τώρα αρχίζει αυτή η προσπάθεια Ελπίζω και εύχομαι να είναι μια καλή βάση το σχέδιο γνωμοδότησης για να κάνετε εσείς προτάσεις και τροπολογίες. Ποια κατεύθυνση θέλουμε να δώσουμε, τι προτεραιότητες έχουμε και ποια είναι τα μελήματά μας. Σταματώ εδώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά θα ακούσω τα σχόλιά σας και τη συνεισφορά σας. Thank you, Vice Chair, for your presentation. And now I would like to give the floor to Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Θα δώσω το λόγο συναδέλφος ο κύριος Πρέντα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου για το ότι σήμερα συζητούμε την αθέρωση των δημοσιονομικών κανόνων που στο το Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης παρά το γεγονός ότι μόνο περίπου και 100 είμαστε Δέκα συνάδελφοι είμαστε μόνο εδώ περίπου και όχι περισσότερο και νομίζω ότι μόνο για 10% μιλάμε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι στην Επιτροπή μας και εγώ ως πρώην εισηγητής για τον προπελισμό της Επιτροπής μας ζητήσαμε πολλές φορές να γίνει αναθεώρηση ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες αυτούς ώστε να προσαρμοστούν προς την σημερινή κατάσταση. Το θέμα της ε, ευελιξίας λοιπόν για τις ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και γρήγοροι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε και πού θα αναζητήσουμε τους απαραίτητους πόρους ώστε να εφαρμόσουμε την μεγαλύτερη ευελιξία. Θα πρέπει να βασιστούμε στα κονδύλια που έχουν ε, ε, οριστεί για τις χώρες ε, τις γειτονικές και για τις υποψήφιες ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αυξήσουμε την ευελιξία και να διασφαλίσουμε το επίπεδο συμμετοχής μας στις χώρες τις γειτονικές. Δεν θα πρέπει να τις θυσιάσουμε κάποιες γειτονικές χώρες χάρη της ε, ευελιξίας. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η θέση μου τουλάχιστον. Επίσης, θα ήθελα πιστήσω την προσοχή σας στα σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου που προβλέπει ότι τα μέτρα που προβλέπονται θα κάνουν πιο πολύπλοκους κανόνες αντί να τους ε, απλουστεύσουν. Δεν θα πρέπει να το παραγνωρίσουμε το σχόλιο αυτό. Ένα δεύτερο θέμα. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, παρούσα κατάσταση, κυρίως όσον αφορά τα καταπιστευτικά ταμεία, τα trust funds. Θα πρέπει να δούμε πριν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο καταστατικό τους, πώς ακριβώς έχει λειτουργεί. Και βεβαίως, πριν να ολοκληρώσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Άντι Κριστέα, για τις τροπολογίες που προτείνει, που πηγαίνουν προς την κατεύθυνση και των δικών μου παρατηρήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέντα, επόμενος ομιλητής, η κυρία Λούζιν. Ja, vielen ähm, ευχαριστώ πολύ. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν διάβασα και τις 250 σελίδες του κανονισμού έτσι μέχρι τελευταίες λεπτομέρειες και δεν τις μελέτησα. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προτάσεις του. Ορισμένες από αυτές μπορούμε να τις υποστηρίξουμε, ας πούμε την ευελιξία ε, στις δαπάνες ε, για την εξωτερική δράση. Συμφωνούμε με την εκτίμησή σας, όπως επίσης και ε, για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των καταπιστευμάτων ως Γκουέντζιέλ ε, μας βρίσκει σύμφωνος και αυτό. Εκφράζουμε όμως κάποιες επικρίσεις γενικότερα ε, προς τα, τα πιστεύματα. Ιδιαίτερα για την ειρήνη στην Αφρική. African Peace Facility, αυτό το ταμείο, προβλέπει χρηματοδότηση στρατιωτικής εκπαίδευσης. Εμείς φρονούμε ότι Καλύτερα να καταργηθεί αυτό το ταμείο. Επίσης, εκφεύγουν του κοινοβουλευτικού ελέγχου αυτά τα καταπιστεύματα. Ε, το λέτε στην τροπολογία 6, αλλά όχι επαρκώς κατά τη γνώμη μας. Και θα κοιτάξουμε μήπως χρειαστεί κάποια πιο συγκεκριμένη τροπολογία. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές αποστολές της ΕΠΑ, εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, αυτό το πολιτικές είναι λίγο παραπλανητικό. Γιατί βασικά αυτό είναι εκπαίδευση χωροφυλάκων. Δεν είναι ακριβώς πολίτες αυτοί. Ούτε τα κονδύλια είναι πολιτικά αμυγός. Αν δεν είναι στρατιωτικές δαπάνες, είναι τουλάχιστον παραστρατιωτικές. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται με την πρόταση αυτή, δεν συμφωνούμε. Μέχρι τις 14 Μαρτίου έχουμε καιρό και θα κάνουμε τις σχετικές μας τροπολογίες. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι Άλλος. Όχι. Λοιπόν, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 14 Μαρτίου, όπως ακούσαμε, 12 η ώρα το μεσημέρι. Στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε μάλλον στις 11 Απριλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ακολουθεί το σημείο 18 στην ημερήσια διάταξη. Ενημέρωση για την αποστολή της ε, Επιτροπή μας αντιπροσωπεία στην Ινδία την περασμένη εβδομάδα 21 με 24 Φεβρουαρίου. Αγαπητοί συναδελφοί, είχαμε μια αποστολή ad hoc στην Ινδία την περασμένη εβδομάδα με έξι μέλη μας, τον κύριο Πρέντα, την κυρία Ζόφκο, Νίνα Γκίλ, ο Γιώ Λάινεν και ο κύριο Ούρμας Πέιτ. Ο κύριος Μπασίε επρόκειται να έρθει μαζί μας, αλλά δεν του, δεν έδωσαν θεώρηση για την Ινδία γέρο στο διαβατήριο του. Και λυπάμαι γι' αυτό το γεγονός. Επίσης το διευκρίνησα και προς τους Ινδούς συνομιλητές μας. Η αποστολή εκεί, το ταξίδι μας ήταν συνέχεια ε, τη Συνόδου Κορυφής Ινδία Ευρωπαϊκής Ένωση, που έγινε πέρσι στα πλαίσια τη στρατηγική εταιρική σχέση που έχουμε με συγκεκριμένο στόχο να εμβαθυνθεί η κοινοβουλευτική διάσταση. Η μόνιμη αντιπροσωπεία που έχουμε για την Ινδία αλλά και η Επιτροπή Εσωτερικού Εμπορίου έστειλαν ε, παράλληλα αντιπροσωπείες στην ε, Ινδία και είχαν και επαφές με διαφόρους συνομιλητές και ομολόγους. Η δική μας επιτροπή νομίζω είχε γόνιμες ε, συζητήσεις στο Νέο Δελχή. Καμιά φορά ήταν και συγκρουσιακές με ε, υψηλούς αξιωματούχους της κυβέρνησης, με το διπλωματικό σώμα, το κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών, καθώς επίσης και αντιπροσώπους και εκπροσώπους ε, ομίλων προβληματισμού, think tank. Δεν έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσει που υποβάλαμε και τα αιτήματα συνεδριάσεων. Παρ' όλα αυτά είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον πρόεδρο τη Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή, τον κύριο Σασι Ταρούα και άλλα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών, τον κύριο Ατζιτούβαλ που είναι σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Άβιντ Παναγκάρια ε, αντιπρόεδρο της ε, Υπηρεσίας Μεταρρυθμίσεων και την κυρία Μανίκα Σάνια Γκάντι που είναι Υπουργός ε, Γυναικών και Παιδιών μεταξύ άλλων. Είδαμε τι συνέχεια δόθηκε στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας του 2016 ασχοληθήκαμε με το διάλογο πολιτικής για θέματα παγκόσμιας και περιφερειακής σημασίας και περιφερειακού ενδιαφέροντος ή ανησυχίας όπως είναι η Ρωσία. Ασφάλεια, σταθερότητα και πολυμερή συνεργασία, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μη διάδοση πυρηνικών όπλων, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καταπολέμηση της πειρατείας και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ αυτών και ε, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Πρέντα θα κάνει έκθεση σχετικά με τα όσα διαπιστώσαμε εκεί για τι πολιτικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ανωσυνδία. Τώρα καταρτίζει την έκθεσή του αυτόν τον καιρό. Στι συζητήσει μα και στη συνέντευξη τύπου ξεκαθαρίσαμε ότι θέλουμε το 2017, φέτος, στο δεύτερο εξάμεινο, να δούμε στην Ινδία νέα διάσκεψη κορυφή, σύνοδο κορυφή μάλλον Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας και θέλουμε πάρα πολύ να προχωρήσουμε τώρα σε ό,τι αφορά τη διμερή Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, την οποία συζητούμε εδώ και πολύ καιρό πλέον. Η επόμενη αποστολή μας θα πάει στο γειτονικό Πακιστάν στις 17 με 21 Απριλίου και βεβαίως όλες οι πολιτικές ομάδες θα ενημερωθούν αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί το ακριβές ε, πρόγραμμα. Αυτά από πλευρά μου. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στους άλλους συμμετέχοντες στην αποστολή αυτή, με πρώτο τον κύριο Χριστιαν Πρέντα. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, πριν από μια εβδομάδα είμαστε στο Δελχή. Και πρέπει να προσθέσω ότι η επίσκεψη ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είχαμε φανταστεί. Και θα πω από την εμπειρία μου ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ότι ήταν η χειρότερη που κάναμε τα τελευταία χρόνια, όπως είπατε κι εσείς, συναντήσαμε τους ε, συναδέλφους ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και ιδιαίτερος ε, τον κύριο Σασίτα Ρου, Τη Βουλής, ε, συναντήσαμε έναν υπουργό. τον υπεύθυνο της σύλληψης των πολιτικών της κυβέρνησης και έναν υπεύθυνο των θεμάτων ασφαλείας σε κυβερνητικό επίπεδο. Αυτά μας ήταν όλα. Δεν μπορέσαμε να συναντήσουμε κάποιο άτομο που να εργάζεται για το Υπουργείο Εξωτερικών. Ούτε τον πρόεδρο της Βουλής, έτσι όπως το είχαμε ζητήσει. Δεν μας δέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πριν από την επίσκεψή μας, Το είχαμε προβλέψει αυτό στο πρόγραμμά μας και το είχαμε συζητήσει το θέμα της επισκέψης αυτής πριν να φύγουμε. Και βεβαίως, όχι γιατί ήταν απόντες όσους θέλαμε να συναντήσουμε, ήταν στην Ινδία. Μια φορά συμβαίνει και συνέβη στο παρελθόν να πάει επισκεφθεί κανείς μια χώρα και ο, ο υπέξ να είναι σε μια συνεδρίαση του ΟΗΕ και δεν μπορεί να αναβάλει το ταξίδι του ή να το αλλάξει αν πρέπει να πάει στον ΟΗΕ, αν είναι ο κύριος Μακάλιστερ και ο κύριος Πρέντα στη χώρα του. Βεβαίως κάποιοι ήταν απασχολημένοι με την προεκλογική εξαρτία, αλλά δεν θέλησαν όμως να μαζευτούν και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το πιστεύω ότι πρέπει να το αναφέρουμε και στην πρεσβεία εδώ διότι νομίζω ότι δεν είναι θετικό αυτό. Από τη στιγμή που θέλουμε να αναπτύξουμε στενότερες σχέσεις με την Ινδία, να μην μας δέχεται κανένας υπεύθυνος από το υπέξ το Ινδικό. Δεν είναι πρόβλημα μη διαθεσιμότητας όπως είπα προηγουμένως ή διότι ήταν απασχολημένοι κάπου αλλού οι κύριοι τους οποίους θέλαμε να δούμε. Και πιστεύω ότι στο μέλλον δεν θα πρέπει να κάνουμε τα ταξίδια αυτά πριν να έχουμε μία σαφή και οριστική επιβεβαίωση ότι θα συναντήσουμε τα άτομα που θέλουμε. Διότι, ε, ε, κοιτάξτε, πολλές φορές χρειάζεται να περιμένουμε μια μέρα ολόκληρη πριν να μας πει κανείς το οτιδήποτε από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από την Βουλή, γιατί αν θα συναντούσαμε τον πρόεδρο της Βουλής Φερρυπίν. Αυτό τώρα από την σκοπιά της τυπικής της επίσημης επίσκεψης. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο της επίσκεψης αυτή, πιο πρακτικά, διαπιστώσαμε πολλούς ενδιασμούς ακόμη και στις συναντήσεις, τις πολύ λίγες συναντήσεις που είχαμε σε σχέση με αυτά που αναμέναμε, πολλούς ενδιασμούς όσον αφορά τη θέση μας, την θέση αρχής που έχουμε. Δηλαδή, ε, το ότι στα πλαίσια της ε, πολιτικής μας, ε, μας μας ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενόχλησε πάρα πολύ τους Ενδού που επισκεφθήκαμε και επισήμω. Και είπαμε και συνέντευξη τύπου ότι και αυτό είναι κάτι όμως το οποίο είναι πασίγνωστο. Τη θέση μας την ε, ξέρουν οι πάντε, Για μας ε, συμβαδίζει πολιτική ε, εξωτερικών σχέσεων και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σε όλες τις συνομιλίες που είχαμε και θέματα στρατηγικών εταίρων, πραγματικά είδαμε ότι τους ενοχλεί το θέμα αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν νομίζω ότι κανένας αγνοεί κάτι το οποίο για μας είναι θεσμικό, αν θέλετε, και πρωταρχικής σημασίας. Όταν μιλούμε, λοιπόν, ε, για εξωτερική πολιτική, μιλούμε με ε, άτομα από τα αντίστοιχα υπέξη και για την πολιτική, την εξωτερικών υποθέσεων και δική μας η Επιτροπή ποτέ δεν διαχωρίζει αυτά που λέγει από την σημασία που προσδίδουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το, αυτό που μας είπαν εν ολίγης ήταν μην ανακατεύεστε σε τέτοιου είδους θέματα. Ήτανε Επίσης πάρα πολύ διαφορετικά που εκφράστηκε και σε θέματα σχέσεων με την Ρωσία και με τη ΣΥΠΑ. Θα πω τώρα δύο λόγια για το πρώτο θέμα, διότι για τους Ινδούς συνομιλητές μας, αυτούς που είδαμε, η σχέση με την Ρωσία και οι κυρώσεις προς τη Ρωσία δημιουργούν πρόβλημα στην Ινδία. Και αυτό το θεωρούν ως ε, έμεση ενθάρρυνση της Ρωσίας να προσεγγίζει περισσότερο την Κίνα. Μεγάλοι λοιπόν ενδιασμοί και εδώ εκφράστηκαν, διότι βλέπουν τη σχέση μεταξύ Πακιστάν και Κίνας ως πάρα πολύ στεχνή, κατά συνέπεια ως ε, επικίνδυνη σχέση για την Ινδία. Και τον επιβάλλονται κυρώσεις προς την Ρωσία γι' αυτό σημαίνει ότι προσεγγίζει η Ρωσία περισσότερο στην Κίνα, πράγμα που σημαίνει ότι δίδεται σημασία και ενέργεια στο Πακιστάν γειτονική τους χώρα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση με την Ινδία. Επαναλαμβάνω, εμείς είπαμε ότι θέλουμε να αναπτύξουμε και είμαστε διαθέσιμοι να έχουμε μία στενότερη σχέση, πιο δυναμική σχέση μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μου όμως δεν μας θεωρούν ως ε, συνομιλητή προτεραιότητας τουλάχιστον σήμερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Στη Γερμανία έχουμε μια παροιμία ε, που λέει το ποτήρι είναι μισό γεμάτο ή μισό άδειο σε όλες τις γλώσσες. Και εγώ προσπάθησα ε, με τρόπο έτσι μάλλον προσεκτικό και διπλωματικό να το παρουσιάσω μισό γεμάτο. Εσείς τα πάτε από τα δόντια για το ίδιο ταξίδι. Μιλάμε για τις ίδιες συνθήκες και για το ίδιο ποτήρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώ Λάινεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Κρίστιαν Πρέντα ε, ασχολήθηκε εντατικά με τα παράπονα που είχε να πει και τα βγάλε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εγώ, για καθυστέρηση στην επιβεβαίωση διαφόρων ραντεβού. Αυτό όμω ήταν ανέκαθεν. Το έχω ξαναζήσει και στο παρελθόν. Δεν είχε να κάνει με τη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία και θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά Τρει αντιπροσωπείες πήγαν την ίδια εβδομάδα στο Δαλχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, πράγμα που σημαίνει και άγχος για τους συνομιλητές εκεί. Οπότε και εγώ θα επιθυμούσα καλύτερο συντονισμό του Κοινοβουλίου των δικών μας ε, αντιπροσωπιών και της αντιπροσωπείας για την Ινδία, που για κάποιους λόγους επέλεξε άλλο δρομολόγιο ε, και άλλο πρόγραμμα από ό,τι θα μας ευόλευε εμάς στην ΑΦΕΤ. Θέλω να αναφέρω κάποια σημεία που και μένα μου έχουν μείνει. Σταμάτησε ο Πρέντα εκεί που ήθελα να αρχίσω εγώ. Εταιρική σχέση, στρατηγική εταιρική σχέση λέμε Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας. Πάντα κάνουμε προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Είχαμε κάποιες συνομιλίες που μας είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοια εταιρική σχέση στρατηγική γιατί δεν έχει ουσία. Είναι γεγονός αυτό. Και έχουμε την εντύπωση ε, και ότι η Ινδία την απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της ασφάλειας εκεί στην περιοχή. και τους απασχολεί τι γίνεται με την Κίνα, τι γίνεται με το Πακιστάν, ανησυχούν γενικότερα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ασφαλείας ε, ακόμα δεν μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Ε, Άρα είναι ε, σημαντικό να πούμε ότι δεν είμαστε στρατηγικός εταίρος ασφαλείας για την Ινδία. Και αυτοί κοιτάνε προς την Αμερική ε, ε, για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει. Αυτό μπορεί να συζητηθεί και ελέγχεται και με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο. Επίσης, εμένα μου έμεινε αυτή η πολύ ισχυρή σύνδεση που έχουν οι ελίτ της χώρας με την Ινδία. Και έχει ε, και παράδοση αυτό και ιστορική. Και τι σημαίνει και η σχέση που έχουν με τον Πούτιν ε, και ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική και για την Ουκρανία. Δηλαδή βοήθεια για την Ουκρανία να μην περιμένουμε από την Ινδία. Επίσης συζητήσαμε και για τον κόσμο αυτό που έχει όλο και περισσότερα αυταρχικά καθεστώτα μέχρι και διδακτορικά ε, συζητήσαμε τι ε, σημασία έχουν τα δημοκρατικά καθεστώτα στον κόσμο. Και εκεί μπορεί να χρειαστεί ένας άξονας Ευρωπαϊκή Ένωση, Ινδία, Ιαπωνία. Δηλαδή να συνεργάζονται δημοκρατικά καθεστώτα απέναντι σε διάφορες προκλήσεις που έχουμε. σε σχέση με ανεξαρτησία του τύπου, της δικαιοσύνης, ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα. Εκεί η Ινδία σίγουρα είναι ενδιαφέρον εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως και να το κάνουμε παραμένει δημοκρατία η χώρα. Αυτά. Τώρα, να βάλω και λίγο νερό στο κρασί μου για τη συζήτηση με τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχαμε εκεί. Τι μας έδειξε, ότι η Ινδία είναι μια χώρα με πολλά πρόσωπα και η σημερινή κυβέρνηση έχει διαφορετική δράση από κάποιες προηγούμενες. Πολύ γρήγορα σε χαρακτηρίζουν ε, ε, αντίπαλο του έθνους. Το διαβάζουμε σε εφημερίδες, δεν ξέρω κάποιο καθηγητή, κάθε μέρα ε, οποιοδήποτε βγαίνει ε, κάποιος και πει κάτι, το χαρακτηρίζουν αντίπαλο του έθνους. Αντινάσιοναλ. Αυτό είναι μια επιθετική έκφραση της κυβέρνησης απέναντι σε διάφορους επικριτές. Και εμεί μιλήσαμε για ελευθερία των ΜΚΟ, για ελευθερία ε, του τύπου. Αυτά έχουν περιοριστεί το τελευταίο διάστημα και το διαπιστώνουμε σε πολλές χώρες. Πακιστάν. Ακούσαμε παράπονα και διαμαρτυρίες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν ε, εκφράζεται αρκετά ρητά, είναι μάλλον επιφυλακτική για την τρομοκρατία που προέρχεται από το Πακιστάν ότι υπάρχουν επιθέσεις τρομοκρατικές και δολοφονικές. Έπρεπε να το ελέγξουμε αν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί μας είπαν ότι δεν τα καταγγέλουμε αυτά. Ε, το Πακιστάν έχει GSP SIN που είναι η Συμφωνία Γενικευμένων Προτιμήσεων SIN και πια τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι και εκεί συζητήσιμα και αφιλεγόμενα ενώ στην Ινδία δεν δίνουμε αυτό το καθεστώς ιδιαίτερα προτιμησιακό. Έχουν και, το, αυτοί το δίκαιο τους. Ε, ε, το Πακιστάν έχει αυτό το καθεστώς του εταίρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ινδία όχι και αν δούμε την κατάσταση των κρατών και τη μετρήσουμε τουλάχιστον ε, μας κάνει εντύπωση αυτή η ανισότητα. Και τελειώνω με αυτό που ε, όλα αυτά τα χρόνια είναι στο επίκεντρο της προσοχής, συμφωνία η εμπορική, νομίζω έχει απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο. Η κυβέρνηση Μόντι ενδιαφέρεται για το Made in India. Θέλει να επενδύσει στην Ινδία και το εμπόριο μαζί μας δεν τους τρελαίνει και πάρα πολύ. Δεν ε, το προωθούν, δεν πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλλον δυστοκία για το επόμενο διάστημα προβλέπω. Ήταν και λίγο ακρότητα μαρτυριασμένη η αποστολή. Δεν πήγαμε στη Βομβάη και μείναν δύο μέρες μόνο. Πάντω είχε αρκετή ουσία για τη συζήτηση και δεν μπορώ να πω ότι ήταν αποτυχία. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ήσασταν καταπληκτικό ε, και Πρόεδρος της αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ αγαπητέ Γιολάινεν για αυτή την εξαιρετική λαμπρή ανάλυση. Πάρα πολύ εύστοχα αυτά που είπατε τα τελευταία. Και εγώ Νομίζω τελικά κινούμαστε προς το μισό άδειο ποτήρι. Υπήρχαν κάποιες επικρίσεις, υπήρχαν κάποια προβλήματα, θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε και να τα λάβουμε ε, υπόψη για μελλοντικά ταξίδια, αλλά όπως είπε ο Γιώ Λάινεν, που είναι πολύ έμπειρος ε, ε, βουλευτής, δεν μπορούμε κάποιες εβδομάδες ή μέρες πριν να κλείνουμε ραντεβού. Και όταν είναι την ίδια εβδομάδα τρεις αντιπροσωπείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Δελχή κυκλοφορούν στην Ινδία, είναι επιπλέον επιβάρεση. Τώρα, επόμενο ο ο κύριο Μπασίρ, που δυστυχώ δεν μπόρεσε να είναι μαζί μα. Γιατί άρχισαν να διεκπαιρεώσουν το αίτημα θεώρηση διαβατηρίου και να του χορηγήσουν κύριο βίζα. Πρόεδρε, πράγματι ήθελα να πάω σε αυτή την αποστολή και απογοητεύτηκα με το θέμα της ε, θεώρησης. Εγώ υποψιαζόμουν ότι δεν θα ερχόταν εγκαίρως η βίζα και σας το είχα πει. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην εκδοθεί. Οι συνάδελφοι στην ομάδα που υπέβαλαν αίτηση μετά από μένα πήραν τη θεώρηση ή δεν τη χρειάζονταν. Εκτός μικροφώνου η συνομιλία με τον κύριο, με τον κύριο Πρέντα. Ξέρω, κάποιες χώρες ε, χρειάζονται βίζα, κάποιες άλλες όχι. Εν πάση το συνεχίστε παρακαλώ. Πράγματι θα συνεχίσω, λέει ο κύριος Μπασίρ. Κάποιοι συνάδελφοι που ήρθαν σε επικοινωνία με την εξοχότητά του Μαντζίπ Σιμπούρη μου είπαν ότι επειδή έχω μιλήσει ανοιχτά για τις καταστρατηγήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ειδική διοικητική ε, διαχείριση του Κασμίρ, αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν μου δόθηκε η βίζα. Είμαι μέλος αυτού του κοινοβουλίου και με πάρα πολλοί στην εκλογική μου περιφέρεια έχουν προέλευση καταγωγή από το Κασμίρ και πρέπει να τους εκπροσωπήσω και να εκφράσω τα συναισθήματά τους. Κάθε εβδομάδα μου ασκούν πιέσεις εμένα που με έχουν εκλέξει λόγω των συνεχιζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κασμίρ. Υπάρχουν σφαιρί, όπλα με σφαιρίδια τύπου πέλετ που χρησιμοποιούν οι αρχές. Έχουν αφήσει πάρα πολλούς πολίτες τυφλούς ή μονόφθαλμους. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκατοντάδες έχουν φυλακιστεί στο Κασμίρ. Κανείς δεν επιτρέπεται να επισκεφθεί το Κασμίρ και αν θέλατε εσείς να πάτε θα σας αρνούνταν οι Ινδικές αρχές την πρόσβαση σε αυτή την επικράτεια. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ζητήσει τη διοργάνωση αποστολή στο Κασμίρ και η Ινδία είπε όχι. Είναι σωστό μια χώρα που θέλει να είναι υποτίθεται ταγός της δημοκρατίας στον κόσμο να μην είναι υπόλογη για τις ε, καταστρατηγήσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως εγώ, εκφράζει αυτές τις απόψεις και θέτει ερωτήσεις για το ε, κατάλογο το, και για τις επιδόσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, θα του αρνούνται τη βίζα τόσο πια ευαίσθητη είναι. Δεν νομίζω. Ούτε θα έπρεπε. Δεν σας ασκώ κριτική που πήγατε. Εγώ θα αρνιόμουν να πάω βέβαια αν είχαν αρνηθεί τη βίζα σε κάποιον άλλον. Το κάνανε επίτηδες συνδικές αρχές ε, σας κράτησαν στο σκοτάδι, σας δώσαν εσάς τις δικές σας βίζες, αλλά δεν σας ενημέρωσαν ότι δεν είχαν κανένα σκοπό να δώσουν σε μένα. Εάν το ξέρατε, είμαι σίγουρος ότι θα είχατε προβάλει αντιρρήσεις και θα το είχατε σκεφτεί άλλη μια φορά του κατά πόσο ε, θα πηγαίνατε ή όχι. Είμαι υπέρ των εμπορικών συμφωνιών με άλλες χώρες, δεν είμαι κατά. Όταν το κάνει όμως αυτό και προβαίνει κανείς σε τέτοιες συμφωνίες, πρέπει να το κάνει με ανθρώπους και με χώρες που έχουν καλές επιδόσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το είπε και ο συνάδελφος, ο κύριος Πρέντα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι στο επίκεντρο Τη διαπραγματεύση πριν τη σύναψη οποιασδήποτε εμπορική συμφωνίας. Και σε αυτή την ανακοίνωση λέγεται ότι ο πρόεδρο τονίζει την ανάγκη για την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του Ειδικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κυρίω μέσω και ιδιαίτερω μέσω αποστολών και επισκέψεων. Αφού τότε αυτό αναφέρεται, δεν θα πρέπει να γίνεται να τρώμε πόρτα ως αντιπροσωπεία και αναφέρεται επίσης Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθεί στο κείμενο ότι μου αρνήθηκαν τη βίζα ειδικέ αρχέ. Θα πρέπει να απεικονίζεται, να αναγράφεται στο κείμενο και να υπάρχει κάποια αναφορά στις ανησυχίες για τι ε, παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρο. σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Υπενθυμίσαμε στους ε, ε, ε, Ινδούς φίλους μας ότι θέλουμε τη δημιουργία μιας ομάδας φιλίας στο Ενδικό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας και θέλουμε να υπάρξει αποστολή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Ειδικού Κοινοβουλίου είναι σε αποστολή. Σε κάθε περίπτωση κύριε Μπασίρ λυπούμαστε βαθύτατα γιατί δεν έγινε έγκαιρη επεξεργασία του αιτήματό σας για βίζα, όποια, ε, όποια και αν είναι οι λόγοι πίσω από αυτό. Ε, δύο ομιλητές, η κυρία Σόφμορ και η κυρία Σκύλ. Γκίλ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ε, διπλωματικές δεξιότητες τις οποίες ξεδιπλώσατε στην αποστολή μας στην Ινδία. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή. γιατί είδαμε τη γεωπολιτική θέση της Ινδίας και τι σημαίνει η Ευρώπη για αυτούς. Ήταν πολύ καλή επίσκεψη, πολύ ενημερωτική. Θέλω να συγχαρώ τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ήταν καλός οικοδοσπότης και έκανε το παν, το καλύτερο που μπορούσε, δεδομένου ότι υπήρχαν τρεις αποστολές ταυτόχρονα. Ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν ασθενής. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Υπηρεσίας για Ευρωπαϊκών Θεμάτων ε, έπρεπε να φύγει επίσης. Σε κάθε περίπτωση είχαμε ενδιαφέρουσες συνομολίες με πρώην πρέσβης ε, και πρώην ε, Υπουργού Εξωτερικών την παραμονή το βράδυ, επικεφαλής της διαμόρφωσης άποψης και πολιτικών τάσεων, μας μίλησαν με πάρα πολύ μεγάλη ειλικρίνεια για τη στρατηγική, για την στρατηγική τους για την ασφάλεια και για τα σχέδια ε, της χώρας αυτής. Συμφωνώ με τον συνάδελφο κύριο Πρέντα. Καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πράγματι να επιμείνει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλό θα ήταν να ακούσουμε και άλλες πλευρές και άλλες αξίες που προβάλλουν άλλοι φορείς. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερη ευαισθητοποίηση, περισσότερη εκπαίδευση, ε, να καταλάβουμε περισσότερο τι σημαίνουν όλα αυτά για αυτούς. Το ανέφεραν κάποιοι συνομιλητές μας στην αποστολή. Νομίζω ότι η αποστολή ήταν πολύ ενημερωτική, πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, πήρε υπόψη της το γεγονός ότι οι προτεραιότητες της Ινδίας δεν είναι ίδιες με τις δικές μας απαραίτητα. Νομίζω ότι αξιοποιήσαμε στο έπακρον ε, το χρόνο της παραμονής μας εκεί. Ε, σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η Ναγκίλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ασκήστε εξαιρετικά την Προεδρία αυτή τη αντιπροσωπεία παρά τα προβλήματα που είχαμε. Πρέπει να πω ότι εγώ ήμουνα σε δύο αντιπροσωπείε και στην ε, και την προσωπία και στη ΣΑΦΕΤ. Και ήταν πολύ θετική η εμπειρία μου. Όπως σας είπα, ήταν ατυχές το ότι δεν μπορέσαμε να συνδυάσουμε κάποιες συναντήσεις, διότι με την Ινδική Αντιπροσωπεία συναντηθήκαμε την πρώτη μέρα με τους υπουργούς, τέσσερις με αυτούς και σε... Πρέπει να πω ότι μεταξύ των τριών αντιπροσωπιών υπήρχαν προγραμματισμένες περίπου 20 συναντήσεις. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπήρχε εσκεμένα πρόβλημα από τη δικιά των, από την μεριά των. Τώρα, εάν δούμε την αντιπροσωπεία της ΑΦΕΤ, συναντήσαμε την αντίστοιχη επιτροπή της Συνδικής Βουλής. Έγινε μία συνάντηση στην οποία όλοι είχαμε κλειθεί, Έγιναν ε, συζητήσεις και γευματίσαμε και μας Τώρα όσον αφορά την κάλυψη από τον τύπο. Ήταν εξαιρετική πρέπει να πω. Ξέρω ότι και ο γενικού περιεχομένου εφημερίδες, ο ηλεκτρονικός τύπος, οικονομικού περιεχομένου εφημερίδες, όλα τα μέσα κάλυψαν πλήρως τις επισκέψεις μας. Καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας για το ότι δεν συναντήσατε τον Πρωθυπουργό. Ήταν όμως απόλυτα σαφές για μας ότι επειδή προβλέπονται εκλογές σημαντικές, δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν αυτές οι συναντήσεις. Τι μάθαμε από αυτές τις συναντήσεις. Πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει να μείνει να πάει κάποιος στην Ινδία ε, και να κάνει την επίσκεψη και στο τέλος να κάνει μια συνέντευξη τυπώχηση στην αρχή. Και στο μέλλον θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι δεν πηγαίνουν τόσες πολλές αντιπροσωπείες μαζί, διότι δεν μπορούν ίσως εκείνοι να καταλάβουν διαφορά μεταξύ των διαφόρων αντιπροσωπείων, πράγμα που δημιούργησε μεγάλη σύγχυση. Δηλαδή, ποιος, ποια αντιπροσωπεία από αυτές που ήταν εκεί, τις τρεις έπρεπε να συναντήσει ποιον. Τώρα, σε σχέση με τα σχόλια του κυρίου Μπασίρ, είναι λυπηρό το ότι καθυστέρησε να του χορηγηθεί η θεώρηση. Ξέρω, εγώ δεν χρειάστηκα βίζα. Άλλοι χρειάζονταν. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι στο παρελθόν οι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν κάνει επίσης σχόλια για το Κασμίρ είδαν να τους χορηγείται ε, θεώρηση και δεν νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι κάποια άρνηση είναι κάτι που στρέφεται προσωπικά εναντίον μας, όπως στην περίπτωση των που είπε ο κύριος Μπασίρ. Κάποια μέλη δεν χρειάστηκε να βγάλουν θεώρηση, ούτε κι εγώ, δεν καταλαβαίνω λοιπόν. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε προς τα θετικά. Εγώ τι μπορώ να σας πω, ότι ήταν αυτά τα οποία μας είπαν οι Ινδοί συναδελφοί ως ε, σχόλια ήταν πιο θερμά, πιο θετικά αν θέλετε, προς όλους εμάς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Δεν θα πρέπει λοιπόν ένα συμβάν ατυχές να επηρεάσει την όλη σχέση μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε θετικοί, να δούμε την σφαιρική εικόνα, την ε, συνολική εικόνα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο θετικά και να φτιάξουμε όλες αυτές τις στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις που θέλουμε. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σόφκο Σιλ για τα θετικά πρόσημα που έδωσαν και ακούσαμε και τις ε, επικρίσεις που έγιναν. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω όλη την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δελή, τους Ινδούς συναδέλφους που μας δέχθηκαν και δικόναν το ταξίδι, την γραμματεία. Σήμερα το πρωί έγιναν κάποιες παρατηρήσεις, τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν θα προετοιμάσουμε την επόμενη επίσκεψή μας στο Πακιστάν. Πιστεύω ότι όπως ελέγχθη σωστά, θα πρέπει να κάνουμε συνέντευξη τύπου στο τέλος της επισκεψής μας και όχι όπως τώρα στην αρχή. Αλλά υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε έτσι όπως έγινε τώρα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση του σημείου αυτού, πράγμα που σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της ομάδας και τώρα θα έχουμε και κλεισμένων των θυρών συνάντηση του Διευρυμένου Προεδρίου